Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Η Ντάφνη Καρουάνα Γκαλιτσία δολοφονήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στη Μάλτα. Με ως ε, θύμα ε, έκρηξης ε, βόμβας αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια ε, απόπειρα, μια εκτέλεση την οποία καταδικάζουμε και ζητάμε κατεπηγόντως ε, ε, καταδίκη των υπετίων η Μάλτα είναι ένα μικρό μέρος όπου όλοι ξέρουν όλους, όπου η Δάφνη αποκάλυψε ε, περιπτώσεις διαφθοράς, τις οποίες και κατέγγειλε στιγνά ε, κατά των πολιτικών ε, Δεν ξέρουμε ποιος ευθύνεται για αυτή την εκτέλεση, για αυτή την δολοφονία και δεν πρόκειται κανένα να καταδικάσουμε χωρίς στοιχεία. Αυτό που είναι ωστόσο βέβαιο είναι ότι η Δάφνη ως ε, μέλος του, της Διεθνούς ε, Ερευνητικής Ομάδας ε, αποκάλυψε και κατέγγειλε τη διαπλοκή πολιτικών εξεχώσεων προσωπικότητων στα έγγραφα του Πάναμα και είχε πολλαπλές πιέσεις δεχτεί. Και αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι χωρίς... έκανε μεγάλες έρευνες στη Μάλτα Η Δάφνη λοιπόν είχε πολλούς εχθρούς, αλλά η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης της άποψης του καθενός αποτελεί, αποτελούν βασικές και θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να την... Να παραπιστούμε. Μαζί με την οικογένεια λοιπόν και τους φίλους της Δάφνης θρυνούμε για αυτή και 20 Φεβρουαρίου του τράχοντος έτους θα την ακούσαμε μαζί με άλλους δημοσιογράφους σε ό,τι αφορά τέτοιες καταγγελίες σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ λοιπόν και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την πρωτοβουλία πολλών πολιτικών ομάδων και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωμέλη στο Στρασβούργο να διοργανωθεί συζήτηση για την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης και ιδιαίτερωση για την Μαλτά. Ζητώ ενός λεπτού συγγύη παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ που τηρήσαμε ενό λεπτού σιγή προ τη της Δάφνης Γαλήσια. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος, δυστυχώ. Excuse me. Ε, Η ειδική κατάσταση για την δολοφονία της Δάφνης οδήγησε τον συνάδελφο Ντέβιτ Κάζη στην κατάθεση Προφορική τροπολογία για την έκθεσή μας. David, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του συναδέλφου. Σα ευχαριστώ για την, αυτή στιγμή, την ιδιαίτερη στιγμή που αφιερώσαμε στην Τάφνη και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εξ ονόματο τη οικογένεια, τη εξ ονόματο της αντιπροσωπεία μου και του κράτου τη Μάλτα για την κατανόηση που δείχνετε σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση. Θα ήθελα να καταθέσω λοιπόν την εξή προφορική τροπολογία, η οποία θα ψηφίσει μετά την 667 ω νέα παράγραφο του σχεδίου έκθεση. Και η προφορική τροπολογία θα είναι ως εξή. Καταδικάζει την δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνη για μία από τι δημοσιογράφου στην πρώτη γραμμή του πυρός για την πόλεμψη της διαφθοράς και του ξεπλήματο χρήματο. και που είχε διερευνήσει εκτενώ ε, το θέμα των γράφων Παναμά και που τηλεφωνήθηκε στι 16 Οκτωβρίου μετά από έκρηξη Βόμβα. Διευκρινίζουμε ότι τέτοιε συνθήκε είναι πραγματικά παράτακτες σε οποιοδήποτε τη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κάζα και θα ήθελα να ζητήσω από την ομάδα να μα διευκρινίσει κατά πόσο συμφωνεί με την ε, τροπολία αυτή. Πρόκειται μια, για μια ουδέτερη, αν θέλετε, προσθέκη συγκεκριμένα για την ταφνα Γκαλίτσια και νομίζω ότι το οφείλουμε στο ίδιο μας το κύρος να προσθέσουμε τέτοιες, ε, τέτοια τροποποίηση. Μάλιστα, να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες για τις δύο εκθέσεις και θα πρέπει να κάνω κάποιες προκαταρτικές παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Σήμερα λοιπόν θα ψηφίσουμε για την έκθεση σχεδίου πρωτοβουλίας και τα σχέδια των συστάσεων με τις ηλεκτρονικές κάρτες μας. Συνολικά 15 γλώσσες έχουμε σήμερα. Έχετε τα έγγραφα τα οποία τα λάβατε μέσα της ομάδας. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις του εισηγητή και των σκιωδών κατέληξαν ε, σε τροπολογίε και αλλαγέ μέχρι και σήμερα το πρωί. Και στι τροπολογίε ε, και στι ε, συμβαστικέ προτάσει είμαστε όλοι οι επαγγελματίε εδώ και ξέρουμε ότι τέτοια πράγματα δυστυχώ σε πολλέ περιπτώσει δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Οι συμβαστικέ προτάσει είναι μόνο στα αγγλικά, οι συντονιστέ και οι σκιώδει και ο εισηγητής, οι εισηγητέ είχαν δύσκολο έργο γιατί συνολικά ξέρετε είχαν 667 τροπολογίες για το σχέδιο πρωτοβουλίας και 783 τροπολογίες για τις συστάσεις. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ο Γεπε Κόφορτ και ο κύριος Γιάτσε και δύο συνεισηγητές ε, ανέλαβαν την βασική πρωτοβουλία για την έκθεση. Οι σκιώδεις ε, συνέβαλα στην κατάρτιση των συμβαστικών προτάσεων και ω εκ τούτου θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να δώσω από ένα λεπτό στους δύο συνεισηγητέ για να μας εξηγήσουν τι ψηφίζουμε σήμερα. Για έχει το λόγο. Thank you so much, Chair. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε καταρχάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλου του συναδέλφους από την Επιτροπή, καθώς και τους σκιώδει ηγητές από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Κάναμε καταπληκτική δουλειά μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό μας, τη γραμματεία και τους υπόλοιπου συνεργάτες μας για το τεράστιο αυτό έργο. Ενώπιον μας τώρα έχουμε μία έκθεση πολύ καλή θα δώσουμε μαζί και με τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε στη συνέχεια ένα πολύ ηχηρό μήνυμα για το ότι είμαστε κατά της ε, διαφυγής φοροαποφυγής και τον αγώνα αυτών ε, δεν θα τον σταματήσουμε, θα τον συνεχίσουμε. Έχουμε σαφείς συστάσεις για το μέλλον, για το τι πρέπει να κάνουμε από κοινού ως κράτη-μέλη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον πολύ σημαντικό αυτό αγώνα, την πολύ σημαντική αυτή μάχη. Και θέλω να πω ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης σήμερα δεν θα σημάνει το τέλος των εργασιών μας, αλλά την απαρχή ε, του έργου μας που έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ τον Γέπε, ο, Πέτ, ο Πίτερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Βέρνερ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω και εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι εργάστηκαν ε, στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής και στη συνεδρία των σκιωδών εισηγητών. Είμαι πεπισμένος πως καταφέραμε τελικά να συντάξουμε πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να τις υποστηρίξουν. Επίσης πιστεύω ότι η σημερινή μέρα αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο της Επιτροπής μας όπως επίσης θεωρώ ότι και οι συστάσεις που έχουμε διατυπώσει είναι ρεαλιστικές και άρτιες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και τώρα μπορεί ο Πρόεδρος να κήρυξει φαντάζομαι την έναρξη της ψηφοφορίας. Yeah, Ναι, συγγνώμη, ξέχασα το μικρόφωνο. Μπορούμε επομένως να ξεκινήσουμε από τους πρασίνους έχω μια αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία και σύμφωνα με τους κανόνες χρειαζόμαστε το 1 πέμπτο των μελών 13 δηλαδή που θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ. Θα πρότεινα λοιπόν να δεχθούμε αυτό το αίτημα των πρασίνων για ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη. Εσείς, οι κομμουνιστές τι είναι, υπέρ, οι σοσιαλδημοκράτες, υπέρ, οι χριστιανοδημοκράτες. Η γκουε φυσικά είναι υπέρ. Ε, φυσικά. Η πράσινη, ναι. Επομένως, και η φιλελεύθερη. Και ο Ντέιβιτ Κόμπερ. <laughs> Ωραία. Επομένως, ε, το λαμβάνουμε αυτό υπόψη και να σας πω επίσης ε, ότι παρά το ότι ήθιστε να γίνετε σε επιτροπές Σήμερα μόνο ε, τα πλήρη μέλη μπορούν να ψηφίσουν. Και τα πραγματικά μπορούν να ψηφίσουν μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι πλήρης, ε, τα πλήρη μέλη, τα τακτικά μέλη. Να κάνουμε λοιπόν ε, μια δοκιμή τώρα για να δούμε πώς είμαστε εδώ. Παρακαλώ να ψηφίσετε. So. Ja, drei Λείπουν τρεις. Εκτός αν δεν θέλετε να ψηφίσετε όλοι, εντάξει. Λοιπόν, 58. Εντάξει, είμαστε με τη την δοκιμαστική ψηφοφορία. Λείπουν δύο. Λείπουν δύο. Εντάξει, τέλος πάντων, μπορούμε να ξεκινήσουμε. με την έκθεση για την έρευνα περιπτώσεων ξεπλήματος χρήματος, φοροποφυγής και φοροδιαφυγής. Τροπολογία 130. Καταρχάς ψήφι υπέρ, κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά, απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβιβαστική υπαριθμόν 1, ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές, μία αποχή, μεγάλη πλειοψηφία είναι υπέρ, γίνεται δεκτή. Πηγαίνουμε στη συμβαστική 2α, ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. 2. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 136. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Ε, εντάξει. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Ε, έχουμε λοιπόν 29 ψήφους υπέρ 26 κατά 3 αποχές. Ε, άρα γίνεται δεκτή 136 και πηγαίνουμε στην 137 ψήφι υπέρ. Το ίδιο θέμα είναι. Στο δικό μου τον κατάλογο η γραμματέα εδώ μου λέει να πηγαίνουμε πάμε στην 138 που είναι η ίδια, ναι. Υπέρ, κατά, αποχές, κατά είναι, αλλά να το ελέγξουμε, 138. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρες. 28 ψήφοι υπέρ, 31 κατά και μία αποχή. Περνάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 140. Ψήφι υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία, εγώ νομίζω πρέπει να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 31 κατά και μία αποχή. Συμβεβαστική 3 τώρα, ψήφι υπέρ. Κατά. 2 είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δύο εποχές. Μία εποχή. Εγκρίνεται τώρα. Τροπολογία 151. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα. Συμβιβαστική υπαριθμών 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. 3 είναι κατά και έχουμε μία αποχή. Ξεχάσαμε μία τροπολογία μου λέτε. Μάλιστα, τροπολογία 153. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. 1.53 ελέγχουμε παρακαλώ. Ε, δεν έχει κλείσει ακόμη ψηφοφορία. Τώρα έχει κλείσει ψηφοφορία. 32 υπέρ, 26 κατά μία αποχή εγκρίνεται. 150. Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική. 6, λέει ο πρόεδρος. 157 πάμε. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι σαφή ο κατάλογο. Πηγαίνουν συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Κάποιες αποχές έχουμε, λίγες ψήφους κατά, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική παριθμόν 7. 157 δεν περιλαμβάνεται. Δύο τμήματα. Εντάξει, ναι, 157 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Όχι. Έχει ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία και μάλιστα σε δύο τμήματα για την 157. Να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. 157 τροπολογία πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας παραπάνω από το έλικα. Ε, λοιπόν, από το ΕΛΚ είναι υπεράριθμο ένα. Εντάξει, το ρυθμίσαμε. Λοιπόν, 27 υπέρ 28 κατά 3 αποχέ. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Υπέρ. Εγκρίνεται δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία. Πηγαίνουμε τώρα στη βαστική ε, την ψηφίσαμε υπέρ. Κατά, στην 7 πάμε. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Dann kommen wir zu Amendment 174. Πάμε στην 174 υπέρ. Κατά. Νομίζω έχει απορριφθεί, αλλά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Όχι ακόμα. 27 υπέρ 30 κατά. Μία αποχή απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Και 8α από κοινού ως προστίκη. 8 και 8α. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υπάρχουν κάποιοι κατά. Τέλο πάντων εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία και τώρα πηγαίνουμε στην τροπολογία 181 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. Συμβιβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Παρακαλώ στο μικρόφωνο να μιλήσετε. Συγγνώμη, έχω και την 183 εγώ. Όχι, καλύπτεται. Καλύπτεται στη συμβιβαστική 9. Α, έχω διαφορετικό κατάλογο, λέει ο κ. Λουκέ. Λοιπόν, συμβιβαστική 9, ψήφι ΠΕΡ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Πηγαίνουμε τώρα στη συμβιβαστική 13, ψήφι ΠΕΡ, Κατά. Αποχές. Δεκτή με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 189 έχουν ζητήσει χωριστή ψηφοφορία στους λιστές δημοκράτες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κατά είναι περισσότεροι, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 24 υπέρ, 35 κατά και μία αποχή. Η 192. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. ίδια πλειοψηφία. Κατά. Απορρίπτεται δηλαδή. 193 και 194 και 195 καταπίπτουν. Πηγαίνουμε... Α, είναι ταυτόσιμες. Μα λένε αν εγκριθεί... Α, μάλιστα. Εντάξει. Επειδή απορρίφθηκε, ναι, πρέπει να ψηφίσουμε την 193, 194 195. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ελέγχουμε, εντάξει, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Περάσα. 25 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Συμβιβαστική 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε στη 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 26 υπέρ, 29 κατά, 4 αποχές απορρίπτεται. 208 ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται μεγάλη διαφορά. 209 ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξω. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν τρεις. Πέρασε ψηφοφορίας. ψηφοφορία. 30 υπέρ 29 κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 210. 210 ψήφι υπέρ. Κατά. Πάλι δεν είναι ξεκάθαρο να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 30 υπέρ 28 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στη 212. Υπέρ. Κατά. Πάλι έλεγχος παρακαλώ αν θέλετε. Έναρξη. Πέρας. 28 υπέρ, 31 ε, κατά, μία αποχή. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε μία φορά ακόμα. Έναρξη. Πέρας. 30 ναι, 28 όχι, μία αποχή εγκρίνεται. Η 16 υπέρ. Κατά. Κατά. Κατά. Και λίγο να σηκώνουμε καλύτερα τα χέρια, παρακαλώ. Για να βλέπουμε καλύτερα. Απορρίπτεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορία. Και πέρας. 29 υπέρ, 29 κατά, δύο αποχές απορρίπτεται. Η 217. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η 218 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 219 υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Δεν ε, ήταν ξεκάθαρο. Το L και υπέρ μάλιστα εγκρίνεται άρα. Σαφές. Περνάμε τώρα στη συμβαστική 22. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές με μεγάλη πλειοψηφία έγκρινεται. 23. Συμβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Οι δύο 25 ταυτόσημοι με την 226. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε, αν και νομίζω ότι απορρίπτεται. Οριακά θα είναι πάντως. Ψηφίζουμε. Τρίτα μία ψήφι υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην 227. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 2.31 παρακαλώ υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 2.33. 2.33. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Οριακό είναι το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 28 ναι, 29 όχι. Απορρίπτεται. Η 2.34 υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ τι ψηφίζει. Απορρίπτεται. Πολύ ωραία. Η 235 ταυτόσιμη με την 238. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δεν είναι σαφής ε, η πλειοψηφία. Ψηφίζουμε. Πέρας. 28 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται ή 236 υπέρ κατά Πάλι ωριακό Ψηφίζουμε. Πέρας. 30 ψηφί υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 2.37. Ε, υπέρ. Κατά. Ίδια η πλειοψηφία νομίζω, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Ψηφίζουμε. Πέρε. 31 η ψηφή, πέρα 28 κατά, εγκρίνεται. Το ίδιο. Η συμβιβαστική 26. πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 239 τώρα σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη. Τέσσερις ψήφοι μας λείπουν. Πέρας. Δύο επιμένουν ότι δεν θέλουν. Ένας. Πέρας. 28 υπέρ, 27 κατά, τρεις αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 245. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Ψεφίζουμε. Πέρας. 31 υπέρ, 25 κατά, 3 αποχές, έγκρινεται. Καταπίπτει 46. 2.47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Άμα θέλετε έλεγχο, έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 33 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Η 2.48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλαχος. Αν και είναι το ίδιο το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι εγκρίνεται. Μάλιστα, πέρασε. 28 υπέρ, 29 κατά και μία αποχή απορρίπτεται. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σεμιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.54. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. 28. Υπέρ. 30. Κατά. απορριβεύεται και μία αποχή. 256 υπέρ. Κατά. Η ίδια η ψηφοφορία. Αποχές. Έλαχος, το. Ψηφίζουμε. Περάσει. 36, 26 υπέρ, 30 κατά απορρίπτεται. 257 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259 υπέρ. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 264. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 262. Υπέρ. Κατά. αφέστε το αποτέλεσμα. Έλεγχος παρακαλώ. Περάσει. 30 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 261. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Ζητώ συγγνώμη. Πέρασε. 28 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται. 263 και 265 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266. 266. Υπέρ. Κατά. Πάλι ωριακό το αποτέλεσμα. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Και πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ 30 κατά. Η 8 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι η ίδια είναι η ισορροπία και η πλειοψηφία, αλλά ας ελέγξουμε. Πέρασε. 29 η ψηφή, υπέρ 30 κατά, καμία αποχή, απορρίπτεται. Η 269. Υπέρ. Κατά. Με μεγάλη πλειοψηφία απορρίπτεται η 267 υπέρ. Οριακό. Οριακός. Ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. είναι ψήφοι υπέρ, 20 είναι κατά, η ψηφία απορρίπτεται. Και η 270 είναι η επόμενη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 71. Υπέρ. Κατά. Ωριακό και πάλι το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε. Πέρας, 30 ψήφι, πέρα 28 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 72. υπέρ κατά πάλι ασαφές το αποτέλεσμα ε, λυπάμαι αλλά είναι όλο οριακές οι ψηφοφορίες θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πέρας ισοψηφία απορρίπτεται η 73. υπέρ Κατά. Αποχές με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. 274. Υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ ψήφισε υπέρ. Υπέρ. Αλλά εγκρίνεται. Ωραία. Η συμβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Τα συνηθισμένα. Ποιο απέχει, κανεί. Α, όχι, μία εποχή. Και τρει ψήφισε κατά. Εντί 78. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία. 79 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Και ένας αρνείται να ψηφίσει. 30 μία ψήφοι υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται. 280 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Οι αποχές. Κάποιες λέγε Εγκρίνεται. Η 281 υπέρ. Υπέρ κατά. Πάλι οριακό το αποτέλεσμα. Ας το ελέγξουμε. Πέρασε. 20 υπέρ, 37 κατά απορρίπτεται με διαφορά. Η 2,2 υπέρ, κατά. Η ίδια αβεβαιότητα με διακατέχει. Ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 31 ψήφοι υπέρ, 27 κατά, μία εποχή εγκρίνεται. Η 283 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Έλεγχο και ζητώ συγγνώμη. Ψηφίζουμε. Περάσουμε. 21 υπέρ, 28 κατά, 2 εποχές εγκρίνεται. 2.40, 84, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. η ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας, ένας αρνείται και η ψηφία. Απορρίπτεται. Η 2.85 παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. ψηφία. απορριπτεται Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 43α και την καινούργια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Η 44α η καινούργια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 290 υπέρ. «290 λέω υπέρ, κατά». Έλεγχος. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το δούμε. Ψηφίζουμε. περάσει ένα ε, δεν ψηφίζει, αλλά δεν είναι και υποχρεωμένο. ισοψηφια Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Ή ε, 291-292. Ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Μάλιστα, έλεγχος. 15 υπέρ, 39 κατά. Σαφές το αποτέλεσμα. Τώρα έχουμε φτάσει εσύ στην 295. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 293. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 48. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται η, 2, η 302 συγγνώμη υπέρ κατά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 302 Πέρας. 28 υπέρ, 28 κρατά, Α, δύο εποχές απαραίτητα. Άμα θέλετε, την επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Αν δεν είναι κανένα αντίθετο, πρόκειται για μία και μόνο τροπολογία, μάλιστα επανάληψη. Υπέρ. Α, όχι, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε. Η 302. 302. Για προσέχετε λίγο παραπάνω όμως. Εκεί στα δεξιά. Η ε, 32 υπέρ 26 κατά. Εγκρίνεται η 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 304 υπέρ. 304 λέω υπέρ. Κατά. Απορρίπτε λέω εγώ, αλλά ας το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε. Τρεις ακόμα να ψηφίσουν. Ένας ακόμα. 23 υπέρ κατά απορρίπτεται. Και περνάμε στην 305. Υπέρ, κατά. Άποχες. Ε, εγκρίνεται. 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 306. Πέρας. από απορρίπτεται. Συμβαστική 53. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 309. Υπέρ. Κατά. Όλο το ίδιο έχουμε. Οριακό το αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε. Πάλι η ισοψηφία απορρίπτεται. 310 και 311 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι. Πέρας. 29 Υπέρ 28 κατά μία εποχή εγκρίνεται. 312. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος και εδώ. Οριακό και μάλιστα ισοψηφία. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 3-16. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. 32 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 3-17. Υπέρ, κατά. Το και ήταν υπέρ. Μάλιστα. Τι λέτε. Εκτός μικροσφόντα σχόλια, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για το μάθημα, λέει ο Πρόεδρος. Εγκρίνεται 3.19 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά έλεγχος Πέρας 30 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται η 20. υπέρ κατά Εγκρίνεται. Η ε, 321 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Τι να σας κάνω. Δεν τα έφτιαξα εγώ έτσι. Άντε άλλοι δύο να ψηφίσουν. Πέρας. 28 υπέρ 28 κατά ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβιβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 327 υπέρ κατά. Να ξαναψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά γιατί πάλι ωριακό το αποτέλεσμα. Αντί 2. Πέρας. 30 υπέρ 26 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 3, 32 παρακαλώ υπέρ. Α, διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφορική τροπολογία. Δεν ήρθαμε σε επαφή με όλες, αλλά με ορισμένες μόνο από τις πολιτικές ομάδες και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η γλώσσα προτείνουμε, τέλος πάντων η διατύπωση που προτείνουμε είναι ότι εκφράζουν τη λύπη τους ότι... Α, δεν είμαστε, στη... δεν είμαστε στην 340. Α, συγγνώμη, είναι μετά. Όχι, είμαστε 333. Ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει πάλι να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. «21 υπέρ 28 κατά». Μία αποχή εγκρίνεται. Τώρα είναι, συγγνώμη, πριν 330, τώρα είναι 333, υπέρ, κατά. Το ίδιο. Ηλεκτρονικά. So, noch einer ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ και το ίδιο και κατά. Τρεις αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 59 με την προφορική τροπολογία. Περβάνς. Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι μαθηματικοί ειδικοί υπολόγισαν ότι για να ψηφίσουμε την έκθεση θέλουμε τέσσερις ώρες. Μήπως σε συμβαστικές να τις ψηφίζουμε διανατά σωστή χειρός και ηλεκτρονικά να ψηφίζουμε τις τροπολογίες για να κερδίσουμε χρόνο. Όχι, Περβάνς, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Γιατί αλλάζουν οι πλειοψηφίες συνεχώς. Για κάθε τροπολογία έχουμε διαφορετική πλειοψηφία. Και με τις συμβαστικές άλλωστε δεν καθυστερούμε. Πάμε γρήγορα. Να τα πω αγγλικά καλύτερα. Λέω, τις συμβιβαστικές να τις ψηφίζουμε διανατάσσως της χειρός και τις τροπολίσεις μεμονωμένες με κατευθείαν ηλεκτρονική ψηφοφορία χωρίς να περνάμε από τη διανατάσσωση της χειρός ψηφοφορία. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορική τροπολογία της Άννα τώρα. Σαν Γκόμες. Ευχαριστώ. Λέει λοιπόν. From 2011 to 2014, European and national banking supervision and national tax authorities were inattentive to capital transfers from Portugal into offshores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 Ε, δωροδόκησε τον ε, Ζωσέ Σόκατα στον πρώην Πρωθυπουργό η Τράπεζα με βάση τις κατηγορίες του Δημόσιου Σαγγελέα, ο οποίος κίνησε και, κίνησε και τη δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν αντιρρήσει. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ με τη συμβιβαστική αυτή όχι. Ο κύριος Λουκέ. Άμα χρειάζεται, ε, μάλλον άμα χρειάζονται τέσσερις ενστάσεις ε, μπορούμε να μην ε, ψηφίσουμε θα έλεγα εγώ αφού έχουμε τέσσερις ενστάσεις γιατί είναι σοβαρές καταγγελίες και είναι μια τροπολογία που σαστικά συνιστά κανονική, είναι τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο. Αν δεν έχουμε καταφέρει να τις παληθέσουμε αυτές τις κατηγορίες, μα ένα σημείο αλλάζει μόνο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το σημείο που αλλάζει. Εγώ κατάλαβα ότι έχουμε ένα τελείως νέο κείμενο εδώ πέρα. Yeah. steht's drin. Τι αλλάζει. The ε, η περίοδο ε, κατά την οποία ήταν υπό την Τρόικα, αυτό διαγράφεται. Δηλαδή, από το 2014 και μετά που λέει η περίοδος οπότε η Πορτογαλία ήταν υπό την Τρόικα και και λοιπά. Είχε χτεθεί εγκαίρος πάντως αυτή η τροπολογία. Okay. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 49 υπέρ 6 κατά 3 αποχές. Εκρίνεται. 342 ψήφι υπέρ. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, ναι. Απευθείας ηλεκτρονικά, όπως είπε υπέρ 342. Λείπει ένας, πέρας. 55 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. 3.43. Άρχεται η ψηφοφορία. Yeah, close. Πέρασε. 6 υπέρ, 50 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. 3.44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 51 ψήφι πέρα, 7 κατά καμία αποχή. Ε, θα είχαμε πάει και πιο γρήγορα μας σκόνα το χέρι, τέλο πάντων. 3.45 ψήφι περ, μάλλον όχι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε, 29 υπέρ, 27 κατά, δύο αποχές εγκρίνεται. 346. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 27 υπέρ 29 κατά. Μία αποχή. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 66. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 352 τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άλλος ένας. 6 υπέρ, 50 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται σαφώς. 353. Άρχεται η ψηφοφορία. Αφού το θέλετε. 5 λείπουν. Παρακαλώ. Τι είπατε. Δεν πρέπει να προσέξω αν λείπουν 10 που δεν έχουν ψηφίσει. Τέλο πάντων, λοιπόν, 28 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. 354. Ψηφίζουμε. Θα ψηφίει 28 όλα. Απορρίπτεται. 355. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. 356. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 υπέρ 26 κατά. Μια αποχή. Εγκρίνεται. 357. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 ήταν κατά και 29 υπέρ, άρα εγκρίνεται. 361, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δύο λείπουν, αλλά κλείνω. 24 υπέρ, 31 κατά και μια αποχή. Απορρίπτεται. 360. Άρχεται. Πέρας. 27 υπέρ 28 κατά. Απορρίπτεται. 362. Άρχεται. Close. Πέρας. 12 υπέρ 42 κατά μια εποχή απορρίπτεται. 364. Άρχεται. Όχι, ξέχασα. 363. Άρχεται η ψηφοφορία. Φαντάζομαι θα εγκριθούμε μεγάλη πλειοψηφία. Πράγμα 46 υπέρ 8 κατά δύο εποχές. Τώρα 364 άρχεται. Πέρας. 2 υπέρ 53 κατά 2 αποχές. Απορρίπτεται. Και με τα χέρια θα το βλέπαμε. Τέλος πάντων. 365. Άρχεται. Close. Πέρασε. 28 υπέρ, 28 κατά. Μια αποχή εγκρίνεται. 366. Άρχεται. Πέρασε. Τριαντιτέσσερις το 21 κατά εγκρίνεται. Από την 367 μόνο το 2, το τμήμα 2 θα ψηφίσουμε. Καλύπτεται το 1. Από την 278 ψήφι υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Έπρεπε να σας πω ότι άρχισε η ψηφοφορία. υπέρ 27 κατά μια αποχή εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην 368. Άρχεται. Πέρας. 28 υπέρ 27 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 369. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 31 υπέρ 25 κατά. Εγκρίνεται. Και μία αποχή είχαμε. 371. Πέρασε. 13 υπέρ 43 κατά μία αποχή. 372-373 είναι ταυτόσιμες. Πέρας. 21 ψηφι 534 τέσσερις κατά μία αποχή. Απορρίπτονται. 370. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 29 υπέρ. 27 κατά εγκρίνεται και μία αποχή. 3.75 έναρξη. Ψη, λήξη. 29 υπέρ 26 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. 3.76 έναρξη. Πέρας. υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. 374 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 28 υπέρ 27 κατά. Μία διαφορά ψήφος εγκρίνεται. 377 άρχεται ψηφοφορία. Υπέρ. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 378. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 46 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. 380. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 382. Πέρας. 26 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 381. Πέρας. 21 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 80 εγκρίνεται. 386 ηλεκτρονικά. Πέρασε. 3 υπέρ 52 κατά 2 αποχές απορρίπτεται. 387 άρχεται. Πέρας. 29 υπέρ 25 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. 388. Ψηφίζουμε. Close. Πέρας. 28 υπέρ 24 κατά 3 αποχές εγκρίνεται. 391. Άρχεται. Να, fehlen noch. Τρεις λείπουν. Κλείνω. 28 υπέρ, 26 κατά, μία εποχή εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 393. Άρχεται. Πέρας. 7 υπέρ, 48 κατά. Μία αποχή. Τι θέλετε παρακαλώ. Η πρόταση της συναδέλφους ε, ε Περβάσε μας έκανε να πάμε λίγο πιο γρήγορα αλλά θα πάμε ακόμα πιο γρήγορα άμα δεν μας διαβάζετε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε μπροστά μας, ε, δεν χρειάζεται να ακούμε. Δηλαδή, ε, πέντε δευτερόλεπτα, ε, αν ε, διαρκούσαν οι ψηφοφορίες και να βάζαμε γρήγορα το δάχτυλό μας στο κουμπί, επίσης πιο γρήγορα θα πηγαίναμε. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να είχαμε λιγότερες χωριστές ψηφοφορίες, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Ξέρω ότι ήταν, δεν γινόταν αλλιώ τέλο πάντων. Και ξέρω και ποιοι το ζήτησαν. Ε, είμαστε τώρα στην 395. Πέρασε. Εγκρίνεται. 396. Πέρας. Εγκρίνεται. 397. Πέρας. Εγκρίνεται. Με πέντε ψηφίες διαφορά. 3,99. 28 υπέρ, 27 κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 400. Κάποιοι λείπουν. Κλείνω. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται με μια ψήφο διαφορά. 403. Πέρας. 28 προς 26. 402. Πέρας. 30 προς 26 εγκρίνεται. 404-405 ταυτόσημες. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 406. Πέρας. 29 προς 25 εγκρίνεται. 407 Δεν έχουν ψηφίσει όλοι. 29 προς 26 εγκρίνεται. 401 όχι. Καταπίπτει. Συμβαστική 88. Υπέρ. Εγκρίνεται. 4.13. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 414. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Οριακά είναι τα αποτελέσματα πάντα. Τρεις δεν θέλουν να ψηφίσουν όμως. 46 υπέρ 7 κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 4-15. Πέρασε. Εγκρίνεται. 416. Πέρασε. Εγκρίνεται με δύο, διαφορά, δύο ψήφους διαφορά. 417. εγκρίνεται με 4 ίους διαφορές 418. Εγκρίνεται με 4 ίους διαφορά 419. Πέρας. 28 προς 27 με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 420. Πέρασε Απορρίπτεται. 421. Πέρας. Απορρίπτεται με μια ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική 97. 97. Υπέρ εγκρίνεται. 425 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται.

Δύο δεν έχουν ψηφίσει ακόμη από αυτούς που έχουν τις κάρτες τους στο μηχάνημα. Πέρας. Απορρίπτεται. 4, 28, 4, 29 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ να ψηφίσετε πιο γρήγορα. Δεν μπορώ να κλείσω την ψηφοφορία αν δεν έχουν ψηφίσει 10. Απορρίπτεται. 4.30. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 431. Απορρίπτεται. 432. 432. τριάντα δύο.

437. Αν προσέχει ο συντονιστής του ΕΛΚ θα πάμε πιο γρήγορα. Συγγνώμη, των σοσιαλδημοκρατών εννοούσα. Απορρίπτεται. 4.38. Θα τα είχαμε ξεκαθαρίσει πιο γρήγορα, τάσω τις χειρός. Απορρίπτεται. 4.33.

Abgelehnt. Απορρίπτεται. 441. Ε, Schließen. Πέρασε. 443 και 444. Ταυτόσιμες.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

Εγκρίνεται. 453. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 448. Λείπουν ακόμη κάποιοι. Απορρίπτεται. 4, 49, 4, 450, συγχωρέστε με. Η 49 κατατέθηκε ξεχωριστά. Η 50. Με μία ψήφα 4, 450. εγκρίνεται με τρία ψήφου, Με τρεις ψήφους. 451. Καταπίπτει. 451. 451. Schließen. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 452.

σκέφτεται. 459. Με δύο ψήφες εγκρίνεται. 460.

Μισοψηφία απορρίπτεται. 467. Συγγνώμη. 464. Με μία ψήφο εγκρίνεται. 467, 468 ταυτόσημες. Απορρίπτεται. 465. Απορρίπτεται. 466. Απορρίπτεται.

Απορρίπτεται. 4,72. Δεν την ψηφίζουμε. Στην επόμενη σελίδα, οι 4,73 και 4,74 είναι αυτόσιμε. Απορρίπτεται. 4,76. με δύο ψήφους διαφορά εγκρίνεται. Συμβαστική 113 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 482. Ηλεκτρονικά. απορρίπτεται. 114 συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έκρινεται. 486 και 487. Ταυτόσιμες. Απορρίπτεται με μεγάλη διαφορά. 4,88. ψηφία. Απορρίπτεται. 491 τώρα. 491. Απορρίπτεται. Συμβαστική 116. Υπέρ. Κατά. Άποχες.

Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 498. Πέρας. Απορρίπτεται. 501. εγκρίνεται 4,99 Πέρασε. Ισοψηφία. Απορρίπτεται άρα. 500. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 503. Και 505 από κοινού. Ταυτόχρονα. Απορρίπτεται. 506. Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 507. Με δύο ψήφους απορρίπτεται. 508. Λείπουν ακόμα κάποιοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 509. Πέρας. Απορρίπτεται. 510. Η συμβαστική 120 υπέρ κατά αποχές με μεγάλη διαφορά εγκρίνεται. 514 ελληνικά παρακαλώ. Η 121 συμβαστική. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 521. Πάλι ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 520. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 522. Πέρας. Απορρίπτεται. 523. Απορρίπτεται. Η 525 σειρά η επόμενη. Η 23 απορριφθήκε. 523. εγκρίθηκε. 526 και 534 ταυτόσημες παρακαλώ. Μία ψήφος διαφορά εγκρίνονται. 527. Πέρας. Πέντε ψήφος διαφορά εγκρίνεται. 528. Ε, Πέρας. Απορρίπτεται δύο ψήφοι διαφορά. 529-535 ταυτόσημες από κοινού. χαράς. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 5.30. Η ισοψηφία απορρίπτεται. 5.31. Πέρας. Εγκρίνεται. 5.32. Πέρας. Απορρίπτεται. 5.33, 5.36. Ταυτόσιμες. Περάς. Με δύο ψήφους απορρίπτεται. 537. Πέρας. Εγκρίθηκε. 538. Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 541. mit ein... Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 124. Υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Και μετά περνάμε λοιπόν στην 593. Ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Συμβιβαστική 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο ψήφοι κατά. Τρεις αποχές. Ε, διαφορά μόνο. 553. Ε, Η 553 παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 555. Λείπουν 6 ψήφοι ακόμα. Περάζει. περίπτωση 556. Πέρας. Εγκρίνεται. 558. Πέρας. Απορρίπτεται. 557. Πέρας. Συμβιβαστική 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 563. Πέρας.

Κάποιοι μας λείπουν ακόμα. Πέρασε. Εγκρίθηκε 566. Πέρας. Εγκρίθηκε. 567. Εγκρίθηκε. 570. Λείπουν ακόμα μερικοί. Πέρας. Εγκρίθηκε. 569. εγκρίθηκε. 572. Μας λείπουν ακόμα κάποιοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Μία ψήφος διαφορά. 573-74. Ταυτόσιμες. Έξι συνάδελφοι ακόμα δεν έχουν ψηφίσει. Είναι οριακά τα αποτελέσματα να ψηφίζετε. Εγκρίθηκε τέσσερις ψήφια διαφορά. 575 τώρα. Εγκρίθηκε συμβημαστική 136. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίθηκε. Ηλεκτρονικά η 584. Απορρίπτεται 585 ηλεκτρονικά. απορρίπτεται. 587 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 586. Πέρας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφου 588. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά 591. Πέρας. Απορρίπτεται. 589. Εγκρίθηκε 589. 590, συγγνώμη. 589. Λείπουν ακόμα μερικοί. Κλείνει όμω η ηλεκτρονική ψηφοφορία και εγκρίθηκε. 592. Απορρίφθηκε η 592. Η 594 τώρα. 594. Μας λείπουν 7 ακόμη. Απορρίπτεται. 596. Εγκρίθηκε. 597 πίπτη, 595. Λείπουν κάμποση ακόμα. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 605. ή ενδιάμεσε καταπίπτουν. Η 605 λοιπόν. Απορρίπτεται. 607. Πέρας. Απορρίπτεται. 606. Η 606 παρακαλώ. Εγκρίνεται. 604. γίνεται με δύο διαφορά 612. Πέρας. Απορρίφθηκε. 615 που είναι ταυτόσιμη με την 616. ψηφίσουν. Πέρας. Απορρίπτονται. 6-19. Απορρίπτεται 6-18. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 627. Απορρίπτεται. 628. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 146. Ψήφι υπέρ. Κατά. Είναι δύο κατά. Αποχές ένας. Εγκρίνεται και πηγαίνουμε στην 642. Υπέρ. Α, όχι, συγγνώμη. Ηλεκτρονικά είναι συγγνώμη. Και πάλι μια ψήφο ήταν η διαφορά. 28 προ 27. Και οι δύο δεν ψήφισαν. Τέλος πάντων. 643. Τρεις δεν έχω ψηφίσει. Πέρασε. Ισοψήφια 28. Απορρίπτεται. 6.45. Πέρας. Δύο ψήφια φορά. Απορρίπτεται. 646. Εγκρίνεται. 648 648-649, ταυτόσημες. Πέρας. Απορρίπτονται. 650. Πέρας. Απορρίπτονται. 651. Πέρας. Εγκρίνεται δύο ψήφι διαφορά. 652. Εγκρίνεται. 653. εγκρίνεται δύο ψήφι διαφορά. 654. Εγκρίνεται. 656. Δύο τμήματα έχουμε, αλλά θα ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο δεν χρειάζεται. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 659. Εδώ έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τους πρασίνους. Λείπουν δύο. 47 υπέρ 10 κατά μία αποχή εγκρίνεται. 661. Να αρχίσει η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Μία ψήφος διαφορά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 153 ψήφι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Ποχές. Δύο. Όχι. Εγκρίνεται. 666. 666 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 667. Εγκρίνεται. Περάμε τώρα στις προφορικές, στην προφορική μάλλον τροπολογία του κύριου Κάζα χρειάζεται να την επαναλάβει, ήδη μας την ανέγνωσε. Δεν χρειάζεται, το άλλους θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, όχι ονομαστικά, απλά σαν επαλήθευση ας πούμε. Στην αρχή μας την παρουσίασε ο κύριος Κάζα. Προφορικά μας την παρουσίασε. Δεν αναφέρονται κόμματα. Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. «56 υπέρ 2 κατά καμία αποχή». Σας ευχαριστούμε πολύ αυτή την τροπολογία. Και όταν εκτυπωθεί θα την διανύμουμε από τη Γραμματεία. Έχουμε τώρα λίγες ακόμη σελίδες τροπολογιών για τις αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε ε, πώς θέλετε. Διανατάσσω στις χειρός. Μπορούμε εδώ. Ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ένα ψήφι περ. Εγκρίνεται. Δύο ψήφι περ. Ηλεκτρονικά τη δύο. Τρεις ψήφοι διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Διανατάσεως παρακαλώ. Δυστυχώς το ίδιο, άρα προχωράμε πάλι με η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 3 άρχεται ψηφοφορία. So, Πέρας, δύο ψήφοι διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 ηλεκτρονικά θα συνεχίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώ. Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Απολύπτεται. Πέντε τροπολογία ηλεκτρονικά. schließen. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Schließen. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 10. Υπέρ. Εντάξει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Εγκρίνεται. 12. Ηλεκτρονικά τη 12. Τρει δεν έχουν ψηφίσει. Μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Δεν είναι σαφές ή ηλεκτρονικά. Αλλά να ψηφίσετε παρακαλώ. Δύο δεν έχουν ψηφίσει και είναι οριακό το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Τέσσερις ψήφοι διαφορά. Τροπολογία 15 ηλεκτρονικά. Άρα ας ψηφίσουμε μάλλον τα χέρια. Τέλος πάντων. Τέλειωσε και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. 16. Ηλεκτρονικά. noch Πέρας. Τέσσερις ψήφοι διαφορά εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Μεγάλη πλειοψηφία υπέρ νομίζω εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Όχι, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε. 5 δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Ή ηλεκτρονικά καλύτερα. Πέντε, εφτά, δεν έχουμε ψηφίσει. Έληξε ψηφοφορία. 28 υπέρ 27 κατά εγκρίνεται. Είναι πάντα πολύ ωραία κατά αποτελέσματα και θέλω παρακαλώ σας παρακαλώ να ψηφίζετε. Τροπολογία 20. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. 29 προς 28 εγκρίνεται. 21 τροπολογία. 21. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερις ψήφοι διαφορά. 22 τροπολογία ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Επτά λείπουν. Έξι, τέλος πάντων κλείνω εγώ τώρα. 28 προς 25 γκρίνεται. Τροπολογία 24. 24. Πέρασε. Εγκρίνεται. 25 τροπολογία. Επτά δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. απορρίπτεται τρεις ψήφοι διαφορά. Συμβιβαστική D, δέλτα, υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 33. Βλέπω ότι παίρνει πιο πολύ, αλλά ούτως ή άλλως ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά, οπότε παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Ναι, 50 υπέρ, 7 κατά, 34. Ψήφι υπέρ. Κατά, κατά είναι περισσότερη, απορρίπτεται. Συμβιβαστική, ε και ε α, ή και α. Ψήφι υπέρ. Κατά, κάποιοι είναι κατά, αποχές, 2, 2 ήταν κατά, εντάξει αποχές συμβιβαστική F υπέρ κατά κάποιοι από ό,τι είδα περισσότεροι όμως υπέρ πηγαίνουμε στην τροπολογία 41 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ή μάλλον όχι ποιοι είναι κατά λέει ο πρόεδρος κατά είναι περισσότεροι άρα απορρίπτεται 42. Υπέρ. Ο, δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 42. Από το ΕΛΚ περισσεύει ένας. Ένας να βγάλει την κάρτα. Μην να μην ψηφίσει. Ωραία. Ευχαριστώ τον ή την συνάδελφο. Τέσσερις ψήφοι διαφορά εγκρίνεται. Και πού είμαστε τώρα? Στο 43. 43 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. ...28 προς 27 Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 45. Και αυτό δεν είναι σαφές να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. Κλείνω τώρα την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στις 46 ηλεκτρονικά. Τρισμένο, Πέρας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 49 τώρα υπέρ. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. «28 όλα» και μια εποχή απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Ηλεκτρονικά. Δύο ακόμη να ψηφίσουν. Δεν είναι και πολύ σαφές το αποτέλεσμα. Τελικά είναι σαφές, απορρίφθηκε. 52. Όχι. 53 Περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 τώρα. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. 10 δεν έχουν ψηφίσει. Εντάξει. Πέραση τη ψηφοφορία. 29 προς 26 εγκρίνεται. Τώρα, συμβιβαστική I, Ι, υπέρ, υπέρ βλέπω, η περισσότερη εγκρίνεται. Τώρα, πηγαίνουμε στην τροπολογία 57 της κυρίας Γκόμης. Ψήφι υπέρ. Κατά. εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά τρεις αποχές ουδής εγκρίνεται και πηγαίνουμε που πηγαίνουμε στην τροπολογία 32 θα ελέγξουμε κατευθείαν Πέρας. Απορρίπτεται. Έξι ψήφι διαφορά. Τροπολογία 67. Διανατάσσος υπέρ, κατά. ΙΣΙΑΡ και φιλελεύθερη και... Είναι σαφές όμως ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Ψήφι υπέρ. Είναι υπέρ, νομίζω, υπέρ. Κατά το ίδιο. Αποχές, άρα εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στη συμβαστική έμμα Μη υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην 77 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 79. Ψήφι υπέρ. Εγκρίνεται. 80 υπέρ, το ίδιο. Εγκρίνεται και αυτή. 81. Δεν είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 82 dafür große mehrheit angenommen 83 εγκρίνεται 83 υπέρ 4 μάλλον κατά απορρίπτεται συμβαστική ο όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πηγαίνουμε στην τροπολογία 127 127 Ναι, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ja, ηλεκτρονικά Okay. Schließen. Πέρας. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. 27 28 Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 27 προς 28. Πηγαίνουμε στη συμβαστική Q. Ψήφι υπέρ. Ψήφε. Κατά. Τρεις. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 102. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Mit 28 äh, Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 103-104 ταυτόσιμες. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Mit Stimmen Mehrheit an. Εγκρίνεται δύο ψήφοι διαφορά. 105. δεν είναι σαφές πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 106. 106 ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Ψήφι υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Υπέρ. Όχι. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Πέντε δεν έχουν ψηφίσει. Πέρασε εγκρίνεται. 111. Δεν είναι σαφές ούτε εδώ. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβιβαστική τι, ταφ. Πέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Μετά, 116. Ψήφι περ, δεν είναι σαφές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. So, schließen. Η ισοψηφία 28 όλα απορρίπτεται. Τώρα, πού πηγαίνουμε. Στην 117. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κάποιος έβαλε την κάρτα του, τι έγινε. 28 προς 27 εγκρίνεται. Κατά πίπτη 118 πηγαίνουμε στην συμβαστική Β. Ψήφι Π. Κατά αποχές, 3 κατά ήταν και αποχές εγκρίνεται. 122 τροπολογία. Ηλεκτρονικά. Πέρες. 29 προς 28 μια αποχή εγκρίνεται. Συμβιβαστική W. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική WA. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το Εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 128. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, δεν είναι σαφές. Ε, λοιπόν, 21 προς 28 και μία αποχή εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία, παρακαλώ. Εσείς, ο συντονιστής. Ναι, εκ μέρους ομάδας του ΕΛΚ. Θέλω να στήσω διακοπή 10 λεπτών. Πέντε λεπτά σας δίνω. Πέντε λεπτά σας δίνω, ναι. Γιατί έχουμε και την επόμενη μετά.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

Κάποιε προκαταρτικέ παρατηρήσει, επιτρέψτε μου. Χτε το βράδυ και σήμερα το πρωί, οι πολιτικέ ομάδε ζήτησαν 170 ε, χωριστέ ε, ψηφοφορίε μετά από 1,5 χρόνο εργασία ε, εδώ στην Επιτροπή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν θα σα πω. Κανονικά, οι πολιτικέ ομάδε θα πρέπει να έχουν καλύτερο συντονισμό. Γι' αυτό λοιπόν υπήρξε και διακοπή από το ΕΛ και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε πριν την τελική ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πού είναι η Ιωνίτα. So, so, wir, Markus, komm. So. So, wir kommen nun zur Schluss. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Ονομαστική ψηφοφορία. Fehlen noch 14. Μας λείπουν ακόμα 14 ψήφοι. Noch 8. 8. Έχουμε κανένα που πρέπει να παρακάτσει. Μήπως στη θέση του τέσσερις ακόμα ψήφοι, λοιπόν. Τέλεια. Μπάλτς. Να παρακαλέσω το εξής. Να παρακαλέσω το εξής. Ο συνάδελφος Πολ Τάγκ ψήφισε. Γιατί δεν είναι εδώ παρόν αλλά ψήφισε. Ο συνάδελφο Πολ Τάγκ. Αυτό απλά να το Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται να ψηφίσει κάποιος που δεν είναι παρόν. Μπορεί κάποιο παρακαλώ να βγάλει την ε, κάρτα του συναδέλφου Πολ Τάγκ. Ιδάλλως ε, θα πρέπει να κάνουμε δημόσια δήλωση εδώ στην αίθουσα ποιο ψηφίζει εξ ονόματο του συναδέλφου του. Δύο ψήφοι μα λείπουν ακόμα παρακαλώ. 57 ψήφισαν. 47 υπέρ 2 κατά 6 αποχές. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. Συνάδελφε Τάγκ, ε, δεν περάσατε απαρατηρητός δεν ήσασταν εδώ παρόν, παρόλα αυτά ψήφιστα ψηφίσατε υπέρ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δίνετε εντολή να ψηφίσει άλλο συνάδελφο. Στη δεύτερη θητεία μου εμ, διώξαμε πρόεδρο επιτροπή. Είναι απάτη αυτή. Δεν ξέρω ποιο ήταν με την καλά τη Μαρίλα Πέν ξεκίνησε καταγγελία και ολόκληρη διαδικασία. Δεν επιτρέπεται. Παρ' όλα αυτά να σας ευχαριστήσω. Ήταν δύσκολο το έργο των εισηγητών, των συνεισηγητών και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο τμήμα. Με μεγάλη και συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι και να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα ελπίζοντας να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα. Ο Σάιμον πρώτος. Τουαλέτα. Τουαλέτα. Ντε. Ένα διαλυματάκι. Κοιτάξτε, πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, δώστε μας πέντε λεπτά για την τουαλέτα. Πρέπει να πάμε τουαλέτα. Oui, ok, ok. Also bitte, Pervenche. Äh, Pervenche, benimm dich jetzt mal und lass hier nicht die Sau raus. I've never been... Pervenche. Πέτρη Σάιμον. Είναι... Ησυχία παρακαλώ, ο Πρόεδρος. Es ist eine wirklich ernst gemeinte Bitte. Der Bericht. Μία σοβαρή έκκληση. Πάλι έχουμε μία έκθεση να ψηφίσουμε με 56 σελίδε και πιο πολλέ συμβαστικέ προτάσει από ό,τι στην προηγούμενη έκθεση άλλη μία ώρα θα χρειαστούμε παραπάνω αν δεν κάνουμε σαφώς πιο γρήγορα και κανείς δεν υποχρεούται εδώ να ψηφίσει. Αν ε, λοιπόν πρόεδρος ε, λέει μετά από 5 δευτερόλεπτα από την έξι ηλεκτρονική ψηφοφορία ότι θα κλείσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ε, α κάνουν τι θέλουν οι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να περιμένει. Όλοι λοιπόν α προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να τελειώσουμε κιόλα. Να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ο πρόεδρο, δεν θα λάβω υπόψη ε, την πρόταση αυτή, αλλά θα ζητήσω το εξή. Αν σε οριακέ αποφάσει 5-6 ε, συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει, δεν είναι δυνατόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όλα όσο πιο σωστά γίνεται, γιατί είναι θέμα των ομάδων μεταξύ του. Οι ομάδε ζήτησαν ψηφοφορίε ξεχωριστέ. Δεν έχω ζητήσει κάτι εγώ. Θα ψηφίσουμε όπω πρέπει λοιπόν. Έναρξη τη ψηφοφορία για το σχέδιο των συστάσεων. Να ξεκινήσουμε με τη συμβαστική 1. Ο συνάδελφος Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ζητήσω από τους συναδέλφους να αναβληθεί η ψηφοφορία επί της συγκεκριμένου φακέλου. Δεν ξέρω για πότε ακριβώς, αλλά υπάρχουν πολλά μέλη της πολιτικής ομάδας που θα φύγουν τώρα διότι έχουν υποχρεώσεις. Δεν είχαμε προγραμματίσει οι περισσότεροι από εμά ότι θα κρατούσε τόσο πολλή ώρα η ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν επιτρέψτε μου ταπεινά να σας θέσω το αίτημά μου για αναβολή της ψηφοφορίας. Όχι, πρόκειται για μια έκκληση του επικεφαλής του ΕΛΚ. Μισό λεπτό, Περβάντς. Εντάξει, μην κάνεις ε? επαναστάσει, λε και δεν ήσουν πέντε χρόνια ε, πρόεδρος της Επιτροπής. Ναι, και για σένα ισχύουν ε, οι κανόνε. Έχουμε λοιπόν αποφασίσει ότι θα έχουμε χρόνο μέχρι τι 5.30. Δεν πρόκειται να το τηρήσουμε. Το θέμα είναι πόσο θα το υπερβούμε το όριο αυτό και δεδομένων των εγγράφων μα. Ε, έχουμε και πάλι πάρα πολλέ ξεχωριστέ ψηφοφορίε. Σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι τι 6 και 4, άμα βιαστούμε κιόλας έχεις το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι είχα αυτή τη φρικτή δουλειά που κάνετε εσείς για 10 χρόνια. Η εμπειρία που έχω είναι ότι η ψηφοφορία αυτή σε δύο τμήματα είναι κάτι το ανήκουστο. Ε, αν πράγματι θα πρέπει να σταματήσουμε τις εργασίες μας πριν από το τέλος των ψηφοφοριών, γιατί ο χρόνος που έχουμε δεν μας επιτρέπει να πάμε μέχρι τέλος, προτείνω να αναβάλουμε, γιατί θα ήταν παράλογο να ψηφίσουμε ένα τμήμα του κειμένου και μετά να σταματήσουμε. Ή να μου πείτε ότι θα πάμε μέχρι το τέλος. Αλλά το να κόψουμε στα δύο τον, τον κατάλογο ψηφοφοριών είναι πάρα πολύ περίεργο. Μάλιστα. What is the proposal? Ποια είναι η πρόταση λοιπόν. Η πρόταση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι η αναβολή της ψηφοφορίας. Το πρώτο τμήμα ε, ψηφίστηκε είναι η έκθεση, το δεύτερο οι συστάσεις. Θα ψηφίσουμε λοιπόν επί της προτάσεως αυτής. Καλούμεθα να ψηφίσουμε. Τώρα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ της πρότασης Ροζάτη και ποιοι είναι κατά. Postpone the Yeah. Forty voters. Only 48. 48 ψηφίσαντες 48 ψηφίσαντες. Τέλος της ψηφοφορίας. 19 υπέρ κατά είναι 30 τη πρόταση. Okay. πρόεδρο μπορώ να λάβω ευθύνη για πολλά πράγματα, αλλά όχι για τον κατάλογο των ψηφοφοριών δεν του έχω προετοιμάσει. Εγώ και ξεκινάμε λοιπόν με τη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφο κατά. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ ειλικρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 29 τροπολογία. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Τριάντα ενα, Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 45. Η 3α, συγγνώμη, συμβιβαστική 3α, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 45. Υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Schließen. Angenommen. Äh, Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Amendment 54. 54. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 55. ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Συμβιβαστική υπαριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 60 ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Εξτένα. Ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 62. Ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 63. Ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 64. Ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Συνδεδαστική έξι. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά εγκρίνεται. Στον κατάλογο των ψηφοφορία έχουμε την 65, η οποία είναι πριν από την συμβαστική 7. Άρα 65 παρακαλώ υπέρ. Μετά, μετά. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Η 65. Λοιπόν, 10 ψήφοι. 8. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 29 ψηφί υπέρ 17 κατά. Τρεις εποχές. Σύμβαστική 7 και 7α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7β. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 80. Ψηφιτροπολογία 80. Ονομαστική κλίση. Δύο ψήφοι μας λείπουν ακόμη. Πέρας. 28 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 81. ηλεκτρονικά. Άλλες ψήφι. Εγκρίνεται. Οκτώ ψήφη υπέρ. Ε, παραπάνω. Ονομαστική κλίση τώρα για την 82. Ψηφίζουμε. με ονομαστική κλίση. Άλλε δύο. Πέρασε. Εγκρίνεται. και οκτώ. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφος ε, κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπερφών 99 υπέρ. Ηλεκτρονικά. Μας λείπουν 7 ψήφοι. Πέρασε. Απορρίπτεται η 100. Επίσης αμφιλεγόμενη και αυτή ηλεκτρονικά θα ελέγξουμε. Με 25 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται. Μία ψήφος διαφορά. 104 και 107 ταυτόσιμες. Ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρα. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 102. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Απορρίπτεται. 120 και 121. Μαζί. Ταυτόσιμες υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 111. 111. Υπέρ. κατά ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά παρακαλώ Und dann kommt 26 äh, zu 25. 26 υπέρ 25 με μία ψήφος με ψήφια ψήφο εγκρίνεται. Και καταπίπτει 115. 117. 117. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά. Ασαφές το αποτέλεσμα. απορρίπτεται. Και τώρα η συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η συμβιβαστική 10, αλλά η 119 θα πρέπει να ψηφιστεί ακόμα ένα μικρό προβληματάκι είχαμε, αλλά ας ψηφίσουμε παρακάτω την 119. Από τη γραμματεία κρέμομαι. Εγώ ό,τι μου πει η γραμματεία. Αφού λέει καταπίπτει. Καταπίπτει. Πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε, λέει ο πρόεδρος, με την 125. Συγγνώμη, συμβαστική υπαριθμών 11. 125, όχι. 125. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά αποχές. Τρεις ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. 131. Χωριστή ψηφοφορία για την το δεύτερο τμήμα. Πρώτο τμήμα, λέει. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Κατά πίπτη. 136. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Η πλειοψηφία εγκρίνεται. 137. Υπέρ. κατά απορρίπτεται. Πιστός υπηρέτης της ομάδας μου. 138. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141. Υπέρ. Ευχαριστώ. Περβάνση. Κατά. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 12 και 12α. Υπέρ. Κατά. David. Εγκρίνεται. 157 και 160 από κοινό ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 158. Και 209 λέει ο κατάλογος μου. Α, όχι, εντάξει. 158 λοιπόν ηλεκτρονικά. Ισοψηφία απορρίπτεται. 29. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται οριακά. 151 και 161 ταυτόσημες. ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Ελεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 174. Ηλεκτρονική επαλήθευση πάλι. Εγκρίνεται. Παρακαλώ να συμμετέχετε όλοι. 175. Ε, Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. εγκρίνεται. 176. μόνο πάλι το αποτέλεσμα. χρονική η χρονικη επαλήθευση. Απορρίπτεται. 177. Επίση αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση. Μισό λεπτό. Εγκρίνεται 179. Έλεγχος. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Δέκα άτομα λοιπόν ακόμη. Πέρας. Εγκρίνεται με τρεις ψήφους ε, διαφορά. 180. Ηλεκτρονική επαλήθευση και εδώ. Επτά ψήφι μας λοιπόν ακόμη. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 182. Και αυτό αμφιλεγόμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 183. Και αυτό αμφιλεγόμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. εγκρίνεται 184 υπέρ κατά απορρίπτεται 185 υπέρ αφιλεγόμενο το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ Άλλοι έξι συνάδελφοι να ψηφίσουν Εγκρίνεται. Συμβαστική 14, υπέρ. Κατά. Μία ψηφο. κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187. Σε τμήματα, με πράσινη. Δεύτερο τμήμα βλέπετε ποιο είναι. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ για το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Α, μόνο το δεύτερο κομμάτι ψηφίζουμε. Δεύτερο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. στην 187. Και τώρα να περάσουμε στην συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Δύο αποχές, μία αποχή. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Για 15α συμβαστική παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Πολλές ψήφοι κατά αλλά σαφώς ε, πιο πολλές οι ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 195, ταυτόσημα με την 196. Χωριστή ψηφοφορία έχουν ζητήσει οι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Υπέρ, ηλεκτρονικά, γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Περάζω. 26 ψήφοι υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Η 203 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 261 υπέρ. Αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση. εγκρίθηκε. Και τώρα φτάσαμε στην 205. Ελεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίθηκε. Η 208. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 206. Αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική. Α, όχι, είναι σαφές. Υπέρ. Κατά. Καταψηφίζεται. Απορρίπτεται. Και τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στη συμβιβαστική υπεριθμό 16. Υπέρ. Πάτα. Εγκρίνεται. 210. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Χωριστή ψηφοφορία. Συγγνώμη, αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα για την επαλήθευση. Εγκρίθηκε. 218. 218 υπέρ για τη 218. Τρεις, τέσσερις. Απορρίπτεται. 219. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορριφθήκε. 220-222 ταυτόσημες από κοινού. Αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέσσερις ψήφοι μα λείπουν ακόμη. Και πέρασε. Εγκρίνεται. 221. ηλεκτρονική επαλήθευση και εδώ. Εγκρίνεται. Η 23 παρακαλώ. Και εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίθηκε. 224. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Με μία εποχή. Συμβιβαστική 18. Υπέρ κατα δυο 2-3 κατά αποχές. Εντάξει. Αποχές, ναι, εντάξει. 2.45. Έξι είναι ταυτόσιμες. Περ. Δεν σαφές ηλεκτρονικά. να ψηφίσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας. Απορρίπτονται. 251. Ηλεκτρονικά. Richtig sehe. Brauchen Zeichen. Απορρίπτεται. 252. Ηλεκτρονικά. Yeah, oui. Ναι, παρακαλώ. Εγώ δεν έχω κάρτα ψηφοφορίας. Θα μπορούσατε ενδεχομένως ε, να δεχτείτε τις ψήφους μου. τάσω χειρός. Όχι. Όχι. Μα έρχεται η κάρτα. Δεν είναι δυνατό σήμερα γιατί έχουμε ξεκινήσει εδώ και δυόμιση ώρες τουλάχιστον τις ψηφοφορίες και χωρίς κάρτα δεν γίνεται να ψηφίσετε. Um έχουμε ξεκινήσει εδώ και δυόμιση ώρες τις ψηφοφορίες. Άρα ζητώ συγγνώμη. Αν έρθει η κάρτα σας... Εσύ δεν είσαι πέρα του να πάμε πιο γρήγορα. Σίγουρα κάποιος θα της φέρει τη συναδέλφου την κάρτα. Εσύ όμως έλεγες να πάμε γρήγορα, Πέτερ. Ε, πρέπει να είσαι συνεπής. Όχι, είναι αντιφατικό. Να περιμένετε ώρες ολόκληρες να ψηφίσουν όλοι σε κάθε ονομαστική και να μην δίνετε τη δυνατότητα τώρα στη συνάδελφο να ψηφεί. Ηρεμήστε αγαπητέ συναδελφό πρόεδρος στις διάφορες ε, ε, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες τουλάχιστον δύο-τρεις συνάδελφοι δεν ψήφισαν και παρόλα αυτά έκλεινα εγώ την ψηφοφορία. Και έχουμε χάσει ως ομάδα, η δική μου ομάδα, όλες τις ψηφοφορίες αυτές. Άρα σας παρακαλώ να είμαστε δίκαιοι εδώ. Λοιπόν, θα έρθει η κάρτα της και τότε θα ψηφίσει συνάδελφος. Νομίζω το ε, έγινε σαφές αυτό. Πού είμαστε τώρα στην 252. Ορίστε που έρχεται και η κάρτα. Ορίστε. Σπαταλήσαμε πέντε λεπτά επειδή δεν είχε την κάρτα η συνάδελφος. 2.52. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ή, μάλλον ψήφι υπέρ. Όχι, δεν είναι σαφές. Ναι, ηλεκτρονικά. Τη 2.52. Τρεις δεν έχουν ψηφίσει. και επειδή δεν είναι το αποτέλεσμα σαφές, είναι προφανές ότι πρέπει να περιμένω. Λοιπόν, απορρίφθηκε. 2.53. Υπέρ, κατά, 5 είναι κατά, ε, αποχές εγκρίνεται. 2.56. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, δεν είναι σαφές. Noch drei? Okay, wir schließen. Εγκρίνεται 26 προς 23. 2.44. Δεν είναι ξεκάθαρο ηλεκτρονικά. Schließen. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 258 και 140 από κοινού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 259. Έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τους πρασίνους. Λείπουν δύο-τρει ακόμη. Λοιπόν, πέρασε ψηφοφορία. 43 υπέρ τα κατά εγκρίθηκε. 2,60. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Angenommen. Εγκρίνεται. 262. Ηλεκτρονικά. Λείπουν δύο. Okay, schließen. Angenommen. Εγκρίνεται. 20 συμβιβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 266-267. Είναι ταυτόσιμες. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Schließen. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά. Είναι κάποιοι κατά, από ό,τι βλέπω, αποχές εγκρίνεται. 2,82. Α, συγγνώμη, συμβαστική 22, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 282. Ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 283. 283. Το ΕΛΚ ε, είναι διχασμένο, δεν ξέρω. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε, εντάξει. I need to sign. Yeah. Okay, noch acht, sechs, die nicht abstimmen. 6 δεν έχουν ψηφίσει. Και ε, πρέπει να περιμένω. Τι να κάνω όταν είναι αμφίρο από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα. Είμαστε στη 284. Και αυτή θα την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Schließen. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,92 υπέρ ή μάλλον καλύτερα ηλεκτρονικά. 293, äh, ja, Λείπουν 6. Πέρασε.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 Από το σχέδιο έκθεσης έχει πέρασει εδώ η 598. Δεν είναι σαφές. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Schließen. Abgelehnt. 599. 599. Ούτε αυτό είναι σαφές. Ψηφίζουμε. Noch vier. Schließen. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 24 συμβιβαστική. Περ, κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 2.98. Ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Και τώρα πηγαίνουμε με ονομαστική ψηφοφορία να ψηφίσουμε το 299. Τη ζήτησαν οι πράσινοι. ονομαστική. Πέντε λείπουν. Is in the voting list. Okay, noch drei. Άλλοι τρεις. Πέρας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στις 301-302. Και αυτό δεν είναι σαφές, οπότε θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Α, εγκρίνεται. 3.15, 17, 3.17. Δεν είναι σαφής. 3.17, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται. Ναι. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο. Δεν ήταν σαφές. Ποιος άλλαξε άποψη. Εγκρίθηκε, δεν εγκρίθηκε. Μα ήταν με μεγάλη διαφορά. 3.18. Ηλεκτρονικά γιατί δεν είναι σαφές. Πέρασε. Εγκρίνονται. 3.20. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά. Viel zu lang diese Liste hier. Noch zwei. Δύο ακόμη. Δεκτή. Ψήφι υπέρ. κατα Σαφώς πολύ κατά. Απορρίπτεται. 324. Ηλεκτρονικά. Πέντε λείπουν. Πέρας. Εγκρίνονται. Κρίνεται. 327. να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 326 καταπίπτει. Μάλιστα. Ναι, ναι, έχει εγκριθεί. Πηγαίνουμε στις 328-329, που είναι ταυτόσιμες. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν έχω ψηφίσει 7 ακόμη. Τέσσερις. Ωραία, πέρασε. Εγκρίνονται. Τα έχω μάθει αυτά από τον Γκουαλτιέρη στην Επιτροπή Έκων. Λοιπόν, συμβιβαστική 27 27. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Από το σχέδιο έκθεση έχουμε είναι 639. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 392. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 349. Ηλεκτρονικά. Μία ψήφος διαφορά εγκρίνεται. Η 350. Περ. Κατά. Απορρίπτεται. 351. Υπέρ. Κατά. Ένας υπέρ, όλοι κατά. Απορρίπτεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 352. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. «24 προς 25 απορρίπτεται με μία ψήφο, διαφορά. 353, 354, 355 ταυτόσημες υπέρ. Κατά απορρίπτονται. 356. Ψήφι υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Danke. Angenommen. Εγκρίνεται. 357. Ελέγχουμε κατευθείαν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, συγγνώμη. Schließen. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30α. Υπέρ. Κατά. εποχές Εγκρίνεται. 358. Ηλεκτρονικά. Fehlen noch 4. Τέσσερις ακόμη. Πέρασε εγκρίνεται. 360. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 361-62. Ταυτόσημες. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 363. Ούτε αυτό είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. Τρεις λείπουν. Πέρας. Απορρίπτεται. 359. Μαμφύρο από το βλέπω. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 ψήφι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32α, ψήφι περ. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 369. Ναι, αμφίρο που είναι ηλεκτρονικά. Noch zwei. okay. Εντάξει, απορρίπτεται. 375-376 ταυτόσημες. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Πού είμαστε? 373. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 373. Τρεις λείπουν. Δέκτη. 374. Όχι. 421. 421. Όχι, όχι. Δεν είναι σαφές ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Abgelehnt. Απορρίπτεται. 374. Δεν σαφές. Ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά. Έξι Έξι δεν έχουν ψηφίσει. Να κλείσουμε την ψηφοφορία. Με μία ψήφο διαφορά απορρίφθηκε. πηγαίνουν στο 379 που και εδώ δεν είναι σε αυτά τα πράγματα. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Angenommen. Δεκτή. 380. δεν μου φαίνεται ξεκάθαρο να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 380. Δέκα δεν έχουν ψηφίσει. Τώρα κλείνω την ψηφοφορία. Δεκτή. 381 τώρα. Ηλεκτρονικά και αυτή. Πέρας. Αδεκτή. Πηγαίνουμε στις 383-384 που είναι ταυτόσιμες. Δεν είναι σαφές, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Οκτώ λείπουν. Απορρίπτονται. 386. Ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε. 387 τώρα ηλεκτρονικά. 387 ηλεκτρονικά. Τρεις να ψηφίσει. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 382. Ηλεκτρονικά. εγκρίθηκε. 385. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ε, εντάξει. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 35 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 398. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 407. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 37. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 408. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 38. Ψήφι υπέρ. Κατά. 2. Αποχές. 1. Εγκρίνεται. Τροπολογία 390 από το σχέδιο έκθεσης. Ψήφι υπέρ. Όχι, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. Άλλοι πέντε λείπουν. Εγκρίθηκε. 422. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 424. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Για τις υποκατηγορίες. 424. Ε, υπέρ, ε, κατά, απορρίπτεται. 425 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές μία και μία κατά. Α, εγκρίνεται. Πού πρέπει να πάω, στην 4.31, όχι. Μετά τη 40. Εγώ αυτή τη σειρά έχω εδώ. Στην 4.31 πηγαίνουμε. Δεν είναι σαφές ηλεκτρονικά. Δεν έχω ψηφίσει 7 ακόμη ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται και περνάμε λοιπόν στη συμβαστική 40 και τότε και μόνο μετά στην 437. Ε, Καταρχάς λοιπόν 14. 40, ε, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται, συμβαστική 40. Και τώρα περνάμε στην 437. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τώρα στην συμβιβαστική 41. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 42. Ή 42 ή 622. 622, τροπολογία 622. Υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 454 445 από πού προήθε ξεχωριστή ψηφοφορία 454 454 Ξεχωριστή ψηφοφορία έχουν ζητήσει πράσινη υπέρ. 454. Αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Εγκρίνεται. 458. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. 460. Κατά. Απορρίπτεται. 462. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. 463. Αμφιλεγόμενο το αποτέλεσμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άλλοι δύο, πέρασε. Εγκρίνεται. 464. Ηλεκτρονικά. Άλλοι τέσσερι ψήφοι. Άλλε τέσσερι ψήφοι. Εγκρίνεται, αλλά πολλοί δεν συμμετείχαν. Συναδελφέ Σίμων. Συμβαστική 44. Υπέρ κατά. Εγκρίνεται. Στο σημείο αυτό, οι διερμηνείς θα σας αποχαιρετήσουν γιατί έχουμε να πάμε σε άλλη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ. Wunderbare Organisation. Ja, wunderbar. Ja.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 480. 480. Controversial. Auf, mach, mach das Ding an. Bitte. Ja, bitte. Okay. Okay. Only 46 members. I miss five.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

Yeah, controversial electronic vote. Ich habe Zeit. Jetzt extra. Nee. I miss three voters. Yeah. Okay, close the vote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 Να. Close. Rejected. 521. Controversial. Five hundred twenty one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

Ten votes. I have a lot of time. We miss five. Okay. Ne, eben waren aber alle da. Adopted. 42.